Τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Σας ενημερώνω ότι έλαβα πολλά αιτήματα για επεξήγηση ψήφου. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 14.45 ε, τα αργότερα για να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες να προετοιμάσουν τη συνεδρίαση για τις 3. Όλες οι επεξηγήσεις ψήφου θα εξεταστούν αύριο μετά από τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Τσούμπερ. Ο κύριος Γκουσκέρι θα μιλήσει εξ ονόματος της ομάδος. για δύο λεπτά παρακαλώ. Γκουσκέρι είναι εδώ. Όχι. Λούαν τότε για ένα λεπτό